ακούει στον κανονισμό του Κοινοβουλίου και συμμετέχει ανάλογα στα όργανα της Ευρωπαϊ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νομική υπηρεσία, η νομική ε, επιτροπή νομικών υποθέσεων στις 11 Ιουλίου επιβεβαίωσε τη κυρία, Ανδρικένε, την εντολή τη κυρία Ανδρικένε και του κυρία Ντοσάντος και πρότεινε λοιπόν ομόφωνα από τις 30 Μαΐου να θεωρούνται ε, εγκεκριμένε οι εντολέ αυτέ. Υπάρχουν αντιρρήσει, όχι. Και άρα λοιπόν ε, επιβεβαιώνεται ο τουρισμό του. Οι αρμόδιε γερμανικέ αρχέ ε, ζήτησαν την άρση τη ακυλία του κ. Γερμαν Βίνκλερ.